Uh, Συνάδελφοι, προτείνω να ξεκινήσουμε. Η σημαντικότερη άλλωστε είναι εδώ. Και προτείνω λοιπόν να αρχίσουμε όπως προβλέπετε από την ημερήσια διάταξή μας με την έκθεση της Μπάρμπαρα Σπινέλη για την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει το λόγο, Μπάρμπαρα. Με ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτά τα λαλάζοντα πλήθη τώρα των βουλευτών, <laughs> χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω το λόγο. Και θα κάνω την παρουσίασή μου στα Ιταλικά. Ευχαριστώ τους κοιόδης εισηγητές την πρόταση έκθεσης ε, την εξέτασαν με μεγάλη προσοχή και συνέβαλαν σημαντικά. Είμαι πεπισμένη ότι σε ορισμένα σημεία θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά και να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς ε, που θα μας βρουν όλου σύμφωνους. Ε, αναφέρομαι σε ζητήματα που αφορούν το ρόλο του οργανισμού θεμελιδών δικαιωμάτων, τη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην εξωτερική δράση της Ένωσης. Κάποιες προτάσεις μου όμως, όπως φαίνεται, δεν χαίρουν συνένεσης από ένα μικρό ή μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών ομάδων. Για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση των εργασιών, ε, για να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε συμβιβαστικές ε, προτάσεις, θέλω σήμερα να υπογραμμίσω μία λογική ε, που με οδήγησε, ε, να σε τη λογική που με οδήγησε σε αυτή την έκθεση, στην ιστορική φάση που ζούμε σήμερα. Δεν ζούμε εύκολες εποχές, ούτε ήρεμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εποχές αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλες ε, διαφωνίες, από διχόνοια, από δυσπιστία προς τα κοινωτικά όργανα. είναι... Είναι μόνο μόνο στις δυσαρέσκειάς μας, όπως λέει ο Σέξπιρ. Εδώ στις Βρυξέλλες ε, εμείς καταλήγουμε να περασπιζόμαστε, έτσι λένε, την παλιά τάξη και είμαστε ανίκανοι να επινοήσουμε μια νέα τάξη. Μας κατηγορούν ε, ότι τα ταμπουρωνόμαστε εδώ ενώ απαιτείται να ακούσουμε περισσότερο τους ανθρώπους και να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις στις ανησυχίες τους. Πολλοί από εσάς ε, ετοιμάζεστε για μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία για την εκλογή του νέου κοινοβουλίου. Το να επανεκκινήσουμε λοιπόν το χάρτη και να του δώσουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες και να διευρύνουμε το πεδίο του θα είναι μια πρώτη απάντηση στη δυσπιστία των ανθρώπων, στο αίτημα για περισσότερα δικαιώματα, στο θυμό που υπάρχει και στη δυσαρέσκεια. Δεν χρειάζεται πια να υπερασπιζόμαστε μια πολιτική τάξη που θρηματίζεται μπροστά στα μάτια μας και να συνεχίζουμε σχέσεις ε, που καταστρέφουν τις πολιτικές ε, και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Να διατηρούμε δηλαδή αυτό που υπάρχει και να απορρίπτουμε οτιδήποτε νέο. Ε, σε συνταγματικά θέματα. Η παλιά τάξη στην οποία αναφέρομαι έχει διάφορες εκφάνσεις, ε, είχε διάφορες εκφάνσεις σε αυτήν εδώ τη θητεία. Πρώτον, η καταστροφή της Ελλάδας. Ο και ο ίδιος, υπενθυμίζω, στις 2 Ιουνίου φέτος ε, μίλησε για την καταστροφή και για την αξιοπρέπεια ενός λαού που καταπατήθηκε λόγω κακή ε, πρόθεση ή αδιαφορία. Η αδιαφορια η πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα του πολιτικού μαζί με το ε, αμάρτημα της παράληψης. Μετά από την Ελλάδα είχαμε το Brexit με κοινωνικές επιπτώσεις πολύ σημαντικές μετά τη σύγκρουση μεταξύ επεκτατικών πολιτικών και πολιτικών λιτότητας ε, όσον αφορά το θέμα του προπολογισμού στην Ιταλία και πιο πρόσφατα τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ε, χρειάζεται να εξετάσουμε κάποια ζητήματα τα οποία αναφέρω εγώ στην έκθεση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και ότι δεν καταλαβαίνουμε και ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με θάρρος και επινοητικότητα κοινωνικά δεινά που οδηγούν στις πολλές αποτυχίες της Ένωσης. Η δυσαρέσκεια των εκλογέων, των ψηφοφόρων, των δικών μας, των δικών σας δεν μπορούμε να απαντάμε με δυσαρέσκεια μιας ε, πολιτικής ε, ελίτ ε, θεσμικής που το μόνο που έχει να δείξει είναι μια διαρκής αδυναμία χωρίς αυτοκριτική και χωρίς να μπορέσει να επανασχεδιάσει την εικόνα της με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά για παράδειγμα τα κοινωνικά δικαιώματα πρώτης προσπαθώντας να διορθώσει τις δυσαρέσκειες, να καταπολεμήσει τον νέο εχθρό, τον λαϊκισμό ε, που απαντά τη δυσαρέσκεια με δυσαρέσκεια και συνεχίζει το χειμώνα αυτό με τον οποίο εμείς ε, ζούμε μέσα στα δεινά χωρίς να πείθουμε τους πολίτες οδηγώντας τους ε, να δείχνουν δυσπιστία και προς το γενικό εκλογικό δικαίωμα. Επειδή δεν υπάρχει σύνταγμα πραγματικό, ξέρετε, το σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκινάει με τις λέξεις «εμείς ο λαός». Και έχουμε το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του δικό μας, ε, της δικής μας ένωσης, όπου η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν η επίση, ότι η επίσημη αναγνώριση της εφαρμογής του οδηγού προενεργά δεν αποτελεί επέκταση των ε, αρμοδιοτήτων της Ένωσης, αλλά πρέπει να αποτελεί την ουσία της. Δεδομένου ότι είναι σχετικά άδεια η αίθουσα, θα μιλήσω για λίγο παραπάνω προσθέτοντας και εξηγώντας κάποια λόγια του Μακεβέλη, ο οποίος λέει ο σοφός ε, λειτουργεί όπως οι τοξότες οι πιο ικανοί, οι οποίοι θεωρώντας ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά και γνωρίζοντας τα όρια του τόξου τους, στοχεύουν πολύ πιο ψηλά από το στόχο. Όχι για να φτάσει το βέλος του σε μεγάλο ύψος, αλλά για να μπορέσουν να φτάσουν στο κέντρο του στόχου ε, χτυπώντας με το βέλος τόσο ψηλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Από το ΕΛΚ, ο Γιώργης Σεφλίν θα μιλήσει εξ ονόματος του Έλμαρ Μπρόκ, όπως και το πρωί άλλωστε. Ευχαριστώ. Ναι, μιλώ εξ ονόματος του Έλμαρ Μπρόκ. Εκείνος βρίσκεται στο συνέδριο του κόμματος στο Βερολίνο. Είναι λοιπόν δικαιολογημένο. Όμως μου άφησε ένα κείμενο το οποίο και θα σας διαβάσω. Βεβαίως ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια Μάρμπαρα για τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο χάρτης αυτός έχει νομική αξία καθώς είναι εισάξιος με τις συνθήκες. Είναι ένα από τα επιτεύγματα της συνθήκης της Λισαβόνας και θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως τέτοιο συχνότερα. Η συγγήτρια έχει κάνει εκτενές έργο μελετώντας την εφαρμογή του χάρτη και έχει καταλήξει και σε μια σειρά από πορίσματα και συστάσεις. Ωστόσο, οι πολλές τροπολογίες που η ομάδα μου έχει καταθέσει σε αυτή την έκθεση δείχνουν ότι η ομάδα μου έχει κάποια προβλήματα με το κείμενο είναι πολλά για να τα αναφέρω ένα προς ένα, αλλά θέλω να εξηγήσω το πρόβλημα που έχουμε με την προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί στην έκθεση αυτή. Γενικά, οι περιορισμοί σχετικά με την εφαρμογή του χάρτη, όπως περιγράφονται στο άρθρο 51, είναι γεγονός που δεν ε, αντικατοπτρίζεται πάντοτε με το σωστό τρόπο στο προτινόμενο κείμενο. Για τα κοινωνικά δικαιώματα, για παράδειγμα, πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι αρμοδιότητε στον τομέα αυτό εναπόκεινται κυρίως στα κράτη-μέλη. Ο χάρτης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις συνθήκες, ούτε να ορίζει καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μπορεί να αλλάζει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που κατοχυρώνονται στις συνθήκες. Ο κίνδυνος είναι ότι αν κανείς αγνοήσει αυτούς τους περιορισμούς μπορεί να δημιουργηθούν φρούδες ελπίδες και προσδοκίες για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ συγγνώμη που δεν θα είμαι σήμερα στην συζήτηση ε, αλλά προσβλέπω στη συνεργασία μας με τους σκιώδεις και θα προσέλθω στις συζητήσεις μας αυτές με επικοδομητικό τρόπο. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο Ραμόν Χάουρεγγι. Δεν είμαι εγώ, αλλά τι να κάνω. Θα μιλήσω εξ ονόματος της συναδέλφου μου, Σίλβια Κάουφμαν. Ε, ε συγγνώμη, ζητεί από την Μπάρμπαρα η κυρία Κάουφμαν η οποία ε, είναι στη Λισαβόνα ε, που έχει συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο ε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω η Πάρβαρα να τη συγχωρέσει. Και θέλω να μιλήσω και εγώ για αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σας πω ότι για την ομάδα μας η έκθεση αυτή ε, της κυρίας Πινέλη είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς ανέκαθεν πιστεύαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε κοινωνική δέσμευση και κοινωνική παρουσία και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. Διότι για ποιο λόγο δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση στις ε, πολιτικές υλοποίησης του κοινωνικού χάρτη είναι επειδή ε, είναι εθνική αρμοδιότητα και αυτό το έχουν διαφυλάξει χώρες και το διατηρούν ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό λείπει αυτή η κοινωνική διάσταση. Ο χάρτης κοινωνικών δικαιωμάτων είναι ε, πλέον πραγματικότητα και ιδιαίτερα μετά την κρίση η κυρία Σπινέλη είχε την ευκαιρία να τα συζητήσει αυτά τα θέματα και εγώ μαζί της ε, σε πολλές εκθέσεις της δικής μας Επιτροπής. Δηλαδή ότι δεν είχαμε μια ανάγνωση έτσι πιο δεσμευμένη και πιο προσιλωμένη στις εντολές του κοινωνικού χάρτη στις διάφορες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράδειγμα, για το μέλλον της Ευρώπης όταν συζητήσαμε έλεγε ότι δεν αντανακλάται ο κοινωνικό χάρτης. Η γεγονό είναι ότι η οικονομική κρίση μας έχει βλάψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια κιόλα. Και μάλιστα έχει βλάψει πάρα πολύ την αποδοχή της κοινωνικής Ευρώπης στα μάτια των πολιτών, που εξακολουθούν ακόμα πολλοί πολίτε να επιθυμούν διακαώ. Και ο κοινωνικό χάρτη μα έχει έτσι ένα ονοδικό χάρτη και η ομάδα μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να βάλει και στην έκθεση αυτή συγκεκριμένα στοιχεία με τις τροπολογίες μας. Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα. Λυπάμαι για την απουσία της Σίλβια, για τους λόγους που σας είπα. Είμαστε στη διάθεση της εισηγήτριας να συνεργαστούμε για μια έκθεση που μας ενδιαφέρει πολύ. Ευχαριστώ. Très bien. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Ραμόν. Οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε απουσιάζουν. Ένα σχόλιο μόνο να κάνω εγώ από πλευρά μου. Εκπλήσωμαι διαβάζοντας αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και συζητώντας με τον Πρόεδρο και με δικαστές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπλήσωμαι από το γεγονός ότι ε, το δικαστήριο θέλει όλο και περισσότερο να βασίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων, που είναι η ε, ανάπτυξη σε λεπτομέρειες των όσων λέει συνοπτικά το άρθρο 2. Εκεί λοιπόν θέλει να βασίζει τις αποφάσεις που εκδίδει το δικαστήριο, γιατί το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τις συνθήκες, να ε, εξακριβώνει, να υπαλληθεύει κατά πόσο οι αρχές, οι θεμελιώδεις αξίες που εγγράφονται στις συνθήκες εφαρμόζονται σωστά στα κράτη-μέλη. Όχι απλώς για λόγους ε, μεταφοράς του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, αλλά και στην εσωτερική ένωμη τάξη της εκάστοτε χώρας και σε ε, τομείς που σε ευρύτατη έκταση μέχρι και 100% είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το δικαστήριο, όχι από εμά, γιατί έχουμε διάκριση των εξουσιών και ε, τη σεβόμαστε και ανεξαρτησία εμείς ε, δεν μπορούμε να προβάλλουμε αντιρρήσεις ή να ενθαρρύνουμε το δικαστήριο προς τη μία την άλλη κατεύθυνση, ούτε έχουμε αντιρρήσεις ε, με τις αποφάσεις. Αλλά να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Ωραία. Κυρία Σπινέλη, θέλετε να επανέλθετε, να απαντήσετε στους ομιλητές. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Φυσικά ευχαριστώ και τον Γιώργη και τον Ραμόν για τις θέσεις των ομάδων τους όπως τις εξέφρασαν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Ραμόν για το διάλογο που ακόμα συνεχίζεται μεταξύ μας και που δεν θα τελειώσει πιθανότατα για το παρόν και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάμε. Προς το παρόν δεν έχω να προσθέσω κάτι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα. Έχουμε λάβει μια εκατοστή τροπολογίες, η προθεσμία έληξε στις 3 Δεκεμβρίου. σήμερα κάναμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες αυτές. Η ψηφοφορία προβλέπεται στην Επιτροπή μας στις 22 Ιανουαρίου, ενώ στην Ολομέλεια δεν έχει ακόμα οριστεί ημερομηνία συζήτησης. Μάλλον Φεβρουάριο ή Μάρτιο, πρώτη δεύτερη σύνοδο του Μαρτίου. Προτείνω τώρα να περάσουμε στο τελευταίο θέμα για την ημερήσια διαταξή μας, η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου είναι γνωμοδότηση ε, προς την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Και στην Επιτροπή Προπολογισμών. Είναι ε, δύο επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας. Δική μας συντάκτη γνωμοδότησης είναι η πρόεδρος μας, Ντανούτα Χιούμπνερ. Και για άλλη μια φορά εκπρόσωπο σήμερα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι ο κύριο Έπφριν που θα μα πει την άποψη τη κύρια Χιούμπνερ. Έχετε το λόγο Γιώργη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μιλώ εξ ονόματος της Ντανούτα Χιούμπνερ. Μου άφησε ένα ε, μακροσκελές κείμενο το οποίο θα σας διαβάσω. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη μεταφορά της ε, συνθήκης ESM σε ευρωπαϊκό δίκαιο και για τη μετατροπή του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα αποτελεί έναν μηχανισμό ε, για τον ε, συμπληρωματικό προς τον μηχανισμό εξυγίανσης. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει το Κοινοβούλιο να δώσει την ε, συγκατάθεσή του. Και όσο ε, ε, εκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου, η ΕΚΟΝ και οι Μπάτζ αποφάσισαν να ε, συντάξουν μια ενδιάμεση έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να τονίσω ότι η ενσωμάτωση των ε, διακυβερνητικών εργαλείων που δημιουργήθηκαν μετά την ε, οικονομική κρίση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ενσωμάτωση αυτή ε, ζητήθηκε επανειλημμένως με εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας. Μεταξύ αυτών την έκθεση για το μέλλον της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Φεβρουάριο του 2017 και την έκθεση Φερχόστατ για πιθανές ε, εξελίσεις και προσαρμογές ε, στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την έκθεση Μπροκ ε, για την βελτίωση για την βελτίωση του θεσμικού πλησίου και τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι η Κομισιόν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα αυτά και κατέληξε σε αυτή την πρόταση για το EMF. Ωστόσο, θέλω να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου για το γεγονό ότι μέχρι στιγμής όλα όσα συζητούνται στο Eurogroup νομικά και πρακτικά αποτελούν μια ε, τροποποίηση της διακυβερνητική συμφωνίας για τον ε, ε, ESM για να εξασφαλιστεί αυτό το backstop. Και παρά το γεγονός ότι η συμφωνία για τον ESM ήταν θετικό βήμα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια μετεξέλιξη ε, είναι ε, ατυχές. Ωστόσο, η έκθεση Μπροκ Μπρέσο ε, ζήτησε την ενσωμάτωση του ESM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπό την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα ελέγχου και παρακολούθησης αυτής της διαδικασίας. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτή η διαδικασία πάντοτε να συνοδεύεται από την κατάλληλη κοινοβουλευτική και δημοκρατική λογοδοσία. Και τώρα, όσον αφορά τα πρακτικά ζητήματα για την εξασφάλιση αυτή τη λογοδοσία και τις τα, προ... τα προαπαιτούμενό τη στην διαφάνεια, θέλω να πω τα εξή. Στην πρόταση τη Κομισιό υπάρχουν διατάξει οι οποίε αποσκοπούν στην εξασφάλιση τη λογοδοσία του EMF στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, το EMF θα πρέπει προφορικό ή γραπτό να απαντά στι ερωτήσει που του απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το EMF θα ε, εκδίδει ετήσια έκθεση η οποία θα διαβεβάζεται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και θα υπάρχει δυνατότητα να οργανώνονται και των θερών συνεδριάσεις ε, με, τον, ε, με τους αντιπροέδρους, τον πρόεδρο και τους ε, εκτελεστικούς διευθυντές του οργανισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό αντικαπτοπτρίζει ακριβώς και τα όσα προβλέπονται για τους άλλους οργανισμούς και τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αρμοδιότητες, το Single Resolution Board, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λειτουργούν εντός του πλαισίου του SSM. Θεωρώ ότι έχουμε μια καλή βάση, είμαστε μια καλή αφετηρία, αλλά θα πρέπει αυτές οι διατάξεις να ισχύουν εξίσου για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και αφού ε, αυτός ο μηχανισμός ολογοδοσίας ε, είναι ε, πολύ τυπικός θα έλεγα δεν θα έλεγα ότι ε, καλωσορίζω ακριβώς ούτε χαιρετίζω την πρόταση της Κομισιόν ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης επίσης θέλω να τονίσω ένα ζήτημα που με ανησυχεί είναι η ανισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην πρόταση για το IMF. E Ενώ το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει έναν μεγάλο κατάλογο αποφάσεων που σχετίζονται με την χορήγηση χρηματοπιστωτικής βοήθειας, οι αλλαγές στο κεφάλαιο του IMF e και άλλα ζητήματα που έχουν δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις, εκεί δεν προβλέπεται ούτε καν κάποια διάταξη ε, μέσω της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωνόταν εγκαίρως για τις ε, αποφάσεις που λαμβάνει το IMF e και εγκρίνονται από το Συμβούλιο θεωρούμε ότι αυτή η ανισορροπία θα, θα δημιουργήσει, ε, μάλλον η, το να ήταν υποχρεωτική η αντίστοιχη διαδικασία και με το Κοινοβούλιο θα ήταν βεβαίω υπερβολικό. Αλλά θέλω τουλάχιστον το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται άμεσα για τις αποφάσεις που λαμβάνει ο ΕΜΕΦ και που εγκρίνονται από το Συμβούλιο. Επίσης, για να μπορεί το ε, Κοινοβούλιο να ε, εκπληρώνει τα καθήκοντά του, οι ε, μηχανισμοί λήψη αποφάσεων θα πρέπει να είναι διαφανείς και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Γι' αυτό και ζητώ ε, υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών σε αυτό το ε, θέμα που θα αντικατοπτρίζεται και στη μελλοντική διοργανική συμφωνία όπως άλλωστε είχε γίνει και στο SSM και στο SRB. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνω ε, από πού προέρχεται αυτή η, ε, αυτό το προαπαιτούμενο το Συμβούλιο να εγκρίνει τις αποφάσεις του EMF ε, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη λήψη αποφάσεων και γι' αυτό ζητώ να υπάρχει σωστή ισορροπία ανάμεσα αφενός στον δημοκρατικό έλεγχο του EMF και τη λογοδοσία του στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και από την άλλη μεριά στην ανάγκη να μπορεί να λαμβάνει τις ε, κατάλληλες αποφάσεις και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έγκαιρα και γρήγορα. Γι' αυτό και ζητώ να γίνει σε βάθος συζήτηση στο Συμβούλιο για, την, ε, για τις διαδικασίες, για την ε, ε, βελτίωση της διαδικασίας κατεπήγοντος ή την δημιουργία ενός άλλου μηχανισμού, το οποίο θα, ο οποίος θα μπορούσε να επιτρέψει την ταχεία λήψη των αποφάσεων με ταυτόχρονη συμμετοχή του Συμβουλίου. Και τέλος υπάρχει και ένα τελευταίο σημείο στην πρόταση που θέλω να επισημάνω και να χαιρετήσω. Το άρθρο 6 για τη λογοδοσία του IMF e e στα Εθνικά Κοινοβούλια των μελών του EMF και άλλων συμμετεχόντων κρατών Υπό την πρόταση της Κομισιόν, το EMF θα πρέπει να διαβιβάζει σε τις εκθέσεις του στα Εθνικά Κοινοβούλια και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτά και προφορικά ερωτήματα στον EMF ή να καλούν τον ε, διευθυντή του EMF για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με την εφαρμογή της, ε, ε, της χρηματοπιστωτικής υποστήριξης. Ε, με δεδομένη λοιπόν τη δομή λήψη αποφάσεων του IMF, ε, είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσει και να έρχονται σε άμεση επαφή. Δημιουργώντα αυτόν τον, ε, το να δημιουργηθεί αυτό ο διάβλο επικοινωνία και λογοδοσία είναι κάτι θετικό. 8 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά μετά τα Χριστούγεννα με τους κοιόδες και όλες τις τροπολογίες που θα καταθέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφα. Ευχαριστήσουμε ε, και την Πρόεδρό μας για την πολύ αναλυτική και εύστοχη σύνοψη της πρότασής της που θα βελτιώσει σημαντικά τα πράγματα και για τις συστάσεις που προτίθεται να κάνει. Η ομάδα των σοσιαλιστών βρίσκεται εδώ, Ραμόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Από τη σκοπιά της δικής μας ομάδας θέλω να πω το εξή. Ευχαριστούμε την κυρία Κιούμπνερ. Ειλικρινά και το Γιώργη, ε, δεν είναι ε, φιλοφρόνηση αυτό, το εννοούμε. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση και ο μηχανισμός αυτός, ε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ε, γίνεται Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Πολύ σημαντικός λοιπόν αυτός ο κανονισμός και ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Υπάρχει ένα εργαλείο, ένα μέσο που μας υποχρέωσε η κρίση να δημιουργήσουμε ε, στην απόλυτη τρικυμία και καταιγίδα των δημοσίων χρεών των διαφόρων κρατών μελών της Ευρωζώνης και παρόλα αυτά ούτε είχε ούτε έχει ε, ένα ε, σωστό θεσμικό πλαίσιο ε, ο μηχανισμός αυτός. Η κυρία Χιούμνερ λοιπόν έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά και συμφωνώ απολύτως και με τη φιλοδοξία της και με την απέτησή της. Η δική μας επιτροπή που έχει την θεσμική, ακόμα και τη συνταγματική ματιά αν θέλετε, για το μηχανισμό αυτό, για το τόσο σημαντικό θεσμό, από την οικονομική και χρηματοπιστωτική σκοπιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει και την υποστήριξη ε, με τη σωστή ε, αρχιτεκτονική, τη θεσμική και την κοινοβουλευτική. Και συμφωνώ απολύτω με την κυρία Χιούμπνερ, γιατί η ΑΦΚΟ οπωσδήποτε, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, θα πρέπει να κάνει τι προτάσει τη στι ε, δύο επιτροπέ που είναι αρμόδιε επί τη ουσία. Η Επιτροπή Προπολογισμών και η Επιτροπή ε, οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων και θα πρέπει να έχει και τη ματιά λοιπόν της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Πρώτον, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το νέο μέσο από τη θεσμική σκοπιά. Αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, έτσι θέλει να το βαφτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. που θα έρθει να καλύψει τα τεράστια ελλείμματα και τα τεράστια προβλήματα που έφερε μαζί του η εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην κρίση μας. Γιατί θα θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι ότι και πάρα πολύ εύλογα και δικαίως υπήρξε πολύ μεγάλη ε, κατακραυγή πολιτική για την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πώς το κάτω-κάτω δεν το επιλέξαμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Εμπλοκή του στη λήψη των αποφάσεων που είχαν τεράστια ε, κοινωνική απήχηση και αντίκτυπο σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης κυρίως, ακριβώς λόγω των ε, συνθήκων και των όρων που βάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η λεγόμενη Τρόικα και συνοδεύεται με την παροχή δανείων ε, στις υπερχρεωμένες χώρες. Χώρες τις οποίες τιμωρούσαν οι αγορές και δεν τις δάνειζαν. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο και εδώ τελειώνει η ιστορία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα ξαναμπεί στην Ευρώπη και πολιτικά αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το τονίζουμε και από τη σκοπιά της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Γιατί τώρα θεσπίζουμε ένα εργαλείο που λέγεται Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Έχει πάνω από 600 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή του για να διασώσει οποιαδήποτε χώρα από μελλοντική κρίση. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτό το νέο εργαλείο, αυτό το νέο μέσο ε, και το αγκαλιάζουμε πάρα πολύ θερμά. Που κατά αυτό αντιστοιχεί στην Ευρώπη που λειτουργεί. Γιατί καμιά φορά όταν μιλάμε για την Ευρώπη που διανύει κρίση και την τιμωρούμε και την ε, κακολογούμε, αλλά όπως έλεγε και ο Ζαμονέα από τις κρίσεις, βγαίνουμε μέρα με τη μέρα, βήμα-βήμα, για να οικοδομούμε το, αυτό το ωραίο αρχιτεκτόνημα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τι λέει η δική μου πολιτική ομάδα για την έκθεση Χιούμπνερ τρία πράγματα που θα προσπαθήσουμε να τις ε, κατασταλάξουμε σε τροπολογίες, γιατί είναι ωραία η έκθεση και φιλόδοξη και πλήρης και απαιτητική, όπως είπα προηγουμένως. Αλλά εμείς έχουμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, θα πρέπει να προσπαθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριλάβει ε, αυτό το θεσμικό όργανο στην ένωμη τάξη και στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Αυτό είναι το πρώτο σημείο της έκθεσης. Αυτό ίσως θα πρέπει να συνοδεύεται και από την εξή σκέψη. Δεν θα είχε νόημα να πούμε από τη δική μας Επιτροπή ότι ε, ένα νέο θεσμικό αρχιτεκτόνημα θα πρέπει να ε, κοσμεί τις νέες συνθήκες μιλάμε για την οικονομική διακυβέρνηση ή της Ευρωζώνης και έχουν δημιουργηθεί διάφορα εργαλεία κατά την ε, πορεία των ετών που θα πρέπει να συμπεριληφθούν με το σωστό τρόπο και να κατοχυρωθούν στις συνθήκες μας. Όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συμπεριλαμβάνει, τα έχει κολλήσει στις ε, κείμενες συνθήκες, αλλά μάλλον θα χρειαστεί κάποια στιγμή να αλλάξουν αυτά. Με ε, προσεχής αναθεωρήσεις των συνθήκων. για να εγγραφούν αυτοί οι σημαντικοί οργανισμοί όπως είναι το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο στις συνθήκες. Από κατά τα άλλα, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ έχω διαβάσει την πρόταση και θέλουν να το βαφτίσουν Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει καλύτερα το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Αλλά στην ΕΚΟΝ μάλλον θα το ονομάσουν αλλιώ. Δεύτερη πρόταση για την έκθεση Χιούμνερ από πλευρά Σοσιαλιστών και Δημοκρατών χρειάζεται να συνδέεται καλύτερα το σύστημα αυτό με την Τραπεζική Ένωση. Γιατί ε, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, στο πούμε έτσι τώρα, θα πρέπει να συνδέεται και να αλληλεπιδρά ως ε, έσχατη καταφυγή χρηματοδότησης όταν έχουμε τραπεζικές κρίσεις. Ακριβώς γιατί ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανση των τραπεζών που είναι και αυτός άλλο εργαλείο που πρέπει να μπει στι συνθήκε και δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να ορίσει ότι μια τράπεζα χρειάζεται ε, χρήματα ε, και για την κεφαλαιοποίηση από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Αυτό δεν το λέει ξεκάθαρα η γνωμοδότηση. Και τρίτον, θα ήθελα το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του να προσθέσει ένα ρόλο στην εκλογή των διευθυντών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Αντίστοιχο με το οργανόγραμμα των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμών της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτά τα τρία έχουμε να προτείνουμε. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ αλλά αυτά έχει να πει η ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Merci, mon cher collègue. Ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Ήθελα να προσθέσω κάποια προσωπικά σχόλια. Όπως είπε πολύ σωστά ο Γεωργή, εξ ονόματος της Ντάρνουτα Χιμπνέρ, Η Επιτροπή ΑΦΚΟ και συνεπώς το Κοινοβούλιο έχει κάνει αυτή την πρόταση επανειλημμένως. Ποιος είναι ο στόχος ε, το να ε, παραμείνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και να μεταμορφωθεί σε ένα πραγματικό εργαλείο όχι πλέον διακρατικό αλλά κοινοτικό. αυτό που εν μέρη προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ικανοποιεί όπως υπόθηκε στο εξή όταν κάποιο κράτος μέλος θα χρειάζεται βοήθεια δεν θα χρειάζεται πλέον να, να τη ζητάμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θα χρειάζεται πλέον να παρεμβαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις ε, ρυθμίσεις ε, και στην παροχή βοήθεια σε ορισμένες χώρες στην Ευρώπη. Ε, κυρίως μέχρι η παρήσφρηση αυτή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν ήταν αποδεκτή από τον κόσμο και ήταν μάλλον αντιπαραγωγική. Πιστεύω ότι πολλοί θα συμφωνήσουμε στο ότι το αρχικό κείμενο της Επιτροπής επιδέχεται κάποιες βελτιώσεις ώστε να εξορροπηθούν καλύτερα οι εξουσίες Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θα πρέπει η διαδικασία να γίνει έτσι ώστε αν ε, παρεμβαίνει το Κοινοβούλιο η διαδικασία να μην ε, καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων διότι όταν μιλάμε για περιόδους ε, οικονομικής κρίσης χρειαζόμαστε γρήγορες διαδικασίες στις οποίες έχουμε ήδη κάποια εμπειρία. Ο Γεωργή υπενθύμησε ότι το SSM και το SRB ως διαδικασίες ε, δίνουν τη δυνατότητα να ληφθούν υπόψη ε, και αυτές οι δύο ανησυχίε με, χωρίς να δημιουργείται κάποια αντίφαση. Κάτι άλλο που πρέπει να αναρωτηθούμε δεν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα τελείω ε, κοινοτικό εργαλείο και να δράσουμε έτσι ώστε τα κονδύλια αυτού του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου να είναι και αυτά κοινοτικά. Να εξηγήσω τι εννοώ. Θα θυμάστε ότι κατά την οικονομική κρίση, η οποία έπληξε πιο πολύ ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημιουργήθηκαν τρία είδη μηχανισμών βάσει της νομοθεσίας που υπήρχε. Πρώτο, είδος μηχανισμού δυνάμενος άρθρο της συνθήκης του οποίου τον αριθμό έχω ξεχάσει αλλά που είναι το ίδιο παλιό με τη συνθήκη της Ρώμης η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή δανείστηκε στις αγορές εξ ονόματος της Ένωσης ώστε να προστρέξει χώρες που δεν ήταν εντός του ευρώ. Το ονομάσαμε ε, βοήθεια ε, για το ισοζύγιο πληρωμών. Ε, αυτό έγινε υπέρ της Ουγγαρίας, της Λετωνίας και της Ρουμανίας. Αυτό εγώ το ονομάζω κοινοτική χρηματοδότηση με κάποιο τρόπο. Τρόπον την δανείστηκε η Ένωση και βοήθησε αυτές τις χώρες οι οποίες επειδή ε, διέτρεχαν δυσκολίες, δεν μπορούσαν να δανειστούν οι ίδιες σε, σε καλές τιμές από τις χρηματαγορές. Βασιζόμενοι λοιπόν ε, ε, στην καλή πίστη της Ένωσης, στην πίστη της Ένωσης, μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί φθηνά για αυτές τις χώρες και τις βοήθησαν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Έχω ξεχάσει και το όνομα και του δεύτερου μηχανισμού που υπήρχε, ο οποίος τι έκανε, εντός της Ευρωζώνης επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί εξ ονόματος ε, της ε, Ένωσης ε, περιορισμένα ποσά νομίζω 60 εκατομμύρια ευρώ 60 δις ευρώ ώστε να, δανείσει, να βοηθήσει χώρες. Δεν θυμάμαι αν ήταν η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία. Και αυτός ο αριθμός που ήταν περίπου 60-70 δισεκατομμύρια υπολογίζονταν από το ΕΚΟΦΗΝ ως δείκτης της ικανότητας δανεισμού της Ένωσης βάσει του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αντιπροσώπευε δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των ανώτων ορίων που ορίζονταν στις δημοσιονομικές προοπτικές και του πραγματικού επίπεδου των ε, πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε κάθε κατηγορία. Ο υπολογισμό αυτός ήταν απόλυτα θεωρητικός. Ωστόσο έγινε δεκτός από τις χρηματαγορές. Αναγνωριζόταν και από τις κυβερνήσεις, ε, το κοινοβούλιο έδωσε ευνοϊκή γνωμοδότηση γεγονός που επέτρεψε στην Κομισιόν να δανειστεί με πολύ χαμηλά επιτόκια ώστε να ε, βοηθήσει αυτά τα κράτη-μέλη που αντιμετώπισαν δυσκολίες. Μαζί παράλληλα με αυτό το ταμείο ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας Αυτός ε, ενισχύθηκε με ποσό 750 δισεκατομμυρίων όπου ουσιαστικά από κοινού χρεώθηκαν όλα τα κράτη της Ευρωζώνης. Δανείστηκαν δηλαδή από κοινού όλα τα κράτη της Ευρωζώνης. Ε, πρόκειται δηλαδή για κάτι διακρατικό, διακυβερνητικό. η ποσοστώσει συμμετοχή, ε, δηλαδή δανεισμού, ώστε να ξαναγίνει επαναδανεισμός, αντιστοιχούσαν ε, στο ε, ΑΕΠ των κρατών μελών. Ο στόχος που θα πρέπει να θέσουμε έχει ως εξής. Το σύνολο των ποσών αυτών εντός του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου θα πρέπει να έχει κοινοτικό χαρακτήρα. Προφανώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ποια είναι η νομική βάση, πώς θα το παρουσιάσουμε νομικά και πόσο, πώς θα το παρουσιάσουμε έτσι ώστε να έχει κάποια οικονομική αξιοπιστία. Όταν μιλάμε για δανεισμό από τις χρηματαγορές, ε, το θέμα της αξιοπιστίας είναι μείζονο σημασία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προκαλέσουμε ανησυχίες στους δανειστές, ε, τους οποίους χρειαζόμαστε. Παρατηρώ όμως ότι έχουμε ένα κανόνα στις συνθήκες, θεμελιώδη κανόνα, από την πρώτη ημέρα της χρηματοδότησης των κοινωτικών πολιτικών, ο ευρωπαϊκός προπολογισμό είναι πάντα ισοσκελισμένος και εκτελείται πάντα ισοσκελισμένος. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Πρόκειται για τον δημόσιο ε, προπολογισμό με την καλύτερη διαχείριση παγκοσμίω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, προπολογισμό στον κόσμο που να μην έχει ποτέ έλλειμμα ούτε μία μέρα το χρόνο. Και σήμερα που είμαστε στις αρχές Δεκεμβρίου είμαστε βέβαιοι ότι ούτε απόψε το βράδυ, καμία μέρα απολύτως, καμία στιγμή δεν υπάρχει έλλειμμα στα ταμεία. Ανά πάσα στιγμή είναι ισοσκελισμένη η εκτέλεση του προπολογισμού. και ο πόρος ε, ε, που σχετίζεται με, το ΑΕΠ, με τα ΑΕΠ έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να αποφεύγεται τέτοιου είδους έλλειμμα. Χάρη σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφού δεν υπάρχει ποτέ έλλειμμα στον προπολογισμό η Ένωση δεν μπορεί να είναι ποτέ χρεωμένη. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει, μπορεί να είναι χρεωμένη και όλος ο κόσμος θεώρησε ότι αυτό ήταν φυσιολογικό μέσω του ισοζυγίου πληρωμών, ε, μέσω του ταμείου αυτού των 60-70 δισεκατομμυρίων που ανέφερα προηγουμένω. Όλα δηλαδή λαμβάνουν χώρα σαν να υπήρχαν δύο ε, λογιστικά, λογιστικοί, ε, λογαριασμοί. Γιατί να μην έχουμε λοιπόν μεγαλύτερο ποσό από 60-70. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε τους διάφορους ειδικού, έχουμε τους διάφορους νομικούς, ε, τους καλύτερους νομικούς τις έχουμε στην ΑΦΚΟ. Ε, να το συζητήσουμε και με όσους ασχολούνται με δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα και εκεί είναι περίπλοκα τα πράγματα. Έχουμε εξαιρετικούς πόρους, ε, εξαιρετικό προσωπικό στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου αλλά θα χρειαστεί να ζητήσουμε και την άποψη συγκεκριμένων εμπειρογνωμόνων. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά ε, σημαντικό, ειδικότερα ε, σε θέματα φιλοσοφίας, ε, κουλτούρας, δόγματος της ΑΦΚΟ, για να αναφέρουμε τέτοιου είδους θεωρίες, να παρουσιάσουμε τέτοιου είδους ιδέες, οι δύο αρμόδιες επιτροπές, η ΕΚΟΝ και η ΜΠΑΤΖ, θα πρέπει να επιδείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Γιώργη δεν θέλει να πάρει το λόγο, ο Ραμόν ούτε αυτός. Πολύ ωραία. Δεν έχω παρά να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, σε περίπτωση που δεν ειδωθούμε. Με κάποιους συνάδελφους θα το ειδωθούμε την επόμενη εβδομάδα. Ε, ίσως όχι τους βοηθούς και τους δερμηνείς και ο Πρόεδρος ε, εύχεται καλές γιορτές ιδιαίτερα τους δερμηνείς. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Διακόπτη συνεδρίαση.